ακάματα συνεχίσει αυτό να το θέτει όποτε βλέπει τις ε, κρατικές αρχές και θα αναζητηθεί έτσι μια λύση. στο πρόβλημα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το Κοινοβούλιο με μεγάλη σαφήνεια ανέφερε την αρχή της αλληλεγγύης που είναι εξαιρετικά σημαντική για μας και χαίρομαι που μας υποστηρίζετε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης που είναι γλώσσες ενός λεπτού. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι η χώρα μου η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο. Πριν δύο μέρες επισκέφτηκε την Ελλάδα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ώρα που ήταν μέσα με τον πρόεδρο της δημοκρατίας ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας δέχτηκε τηλεφώνημα από την κυρία μέρκελ που τον συμβούλευε μαζί με τις εκλογές να γίνει δημοψήφισμα αν ο ελληνικός λαός δέχεται τα μέτρα του μνημονίου ή αν θέλει να φύγει από το euro. ο κύριος ε, σουλτς είδε την οργή είδε την ανεπιφύλακτη καταδίκη τέτοιων παρεμβάσεων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. παρ' όλα αυτά κύριε πρόεδρε ενώ θα περίμενε κανείς αντί να έρχεται και να προπαγανδίζει θέσεις τις οποίες έχει απορρίψει ο ελληνικός λαός να έκανε δήλωση τη δημοκρατική δήλωση που είχε καθήκον ότι θα πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστος ο ελληνικός λαός να αποφασίσει δημοκρατικά δεν το έκανε. τέτοιες συμπεριφορές τέτοιες παρεμβάσεις πλήττουν τη συνοχή της ευρωπαϊκής ένωσης πλήττουν τη δημοκρατία όχι μόνο στην ελλάδα αλλά και στην ευρωπαϊκή ένωση και περιμένω τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να τοποθετηθεί σύμφωνα με αυτή τη δημοκρατική αρχή. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. <coughs> Mr. President, colleagues. we all Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε όλοι μάρτυρες της εργασίας και είδατε ότι ακυρώνονται σημεία από την συνδιάσκεψη των Προέδρων. Υπήρχε ένα ψήφισμα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν και βάσει ποιου κανόνος το κείμενο αυτό το οποίο έχει υιοθετηθεί ξαφνικά άλλαξε η θέση του στην ημερήσια διάταξη και αυτό έγινε από αφόρπαση που δεν ελήφθη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο λόγω κάποιων γλωσσικών σφαλμάτων που ανακαλύφθηκαν στο κείμενο μετά την ψηφοφορία. Διορθώθηκαν όμως τα σφάλματα αυτά και μοιράστηκαν και θεωρούμε ότι δεν δικαιολογείται μία τέτοιου είδους ε, ε, αλλαγή από τη στιγμή που αυτό το ψήφισμα είχε ψηφιστεί και εγκριθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούρτες Λάστρα. Ε, Derek Wokan következik. Δεν είναι παρόν. Derek Wan. Thank you, uh, President. Uh, I speak to welcome the... Νομίζω. Σχετικά με το ταμείο αυτό το οποίο προτείνεται Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα υποδομών στην Ευρώπη τα οποία είναι ικανά να οδηγήσουν την Ευρώπη στην ανάπτυξη. Οι επενδύσεις αυτές οι κοινοτικέ είναι απαραίτητες και στη δική μου περιοχή, στη χώρα μου, στην Ουαλία υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών. Εξηλεκτρισμός σαν παράδειγμα του δικτύου του σιωδρομικού που συνδέει τη Δυτική Ουαλία με το Λονδίνο η τοπική κυβέρνηση προτείνει την ηλεκτροδότηση μόνο μέχρι το Κάρντιφ ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να χρηματοδοτηθεί μέχρι το Σουόνσι. Αυτό είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα δώσουμε τη δυνατότητα και στην Ουαλική κυβέρνηση να δημιουργήσει μία πρόταση, να κάνει μία πρόταση για τη σωστή χρήση των κοινοτικών ταμείων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Ευχαριστώ Στην χώρα των Βάσκων, το Eurobask στις 9 Μαΐου ενέκρινε κείμενο, ένα μανιφέστο και είπαμε οι φιλοευρωπαίοι Βάσκοι ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας στη φιλοευρωπαϊκή γιατί χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα βάλει τον πολίτη στο κέντρο αυτής της ολοκλήρωσης και όχι την αγορά στο κέντρο της ολοκλήρωσης χρειάζεται ένα, ε, μια αναλλακτική πρόταση για την παγκοσμιοποίηση να έχουμε πολυμερείς φορείς και έτσι να ελέγχονται οι χρηματαγορές θέλουμε επομένω μια διακυβέρνηση ευρωπαϊκή και έτσι να βοηθά την οικονομία και η οικονομία να δημιουργεί κοινωνική ευημερία. Και να μην ε, έχουμε, για μια οικονομία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρα, πέρα από, το, από, την, από το χρέος. Χρειάζεται να φτιάξουμε απασχόληση, χρειαζόμαστε μηχανισμούς συνοχής, περισσότερο διάλογο, περισσότερη εξωτερική πολιτική και θέλουμε ένα κατηγορηματικό όχι προς αυτούς οι οποίοι δαιμονοποιούν τους μετανάστες και τις μειονότητες και οπότε έτσι τελικά θέλουμε μια νέα Ευρώπη μια νέα Ευρώπη η οποία να είναι ένα παράδειγμα προς μί, μίμηση να είναι δίκαιη αυτή η Ευρώπη και να είναι χρήσιμη Σας ευχαριστώ Ο επόμενος ομιλητής είναι Ο Νίκος Γρηγολέγος από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί η δημοσιονομική κρίση εφαρμόζονται μέτρα που ξεσηκώνουν την αντίδραση της κοινωνίας ενώ θα μπορούσε να έχει προωθεί μια πολιτική που θα είναι κοινωνικά πιο ισορροπημένη. Αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται καθόλου μέσα στο νέο μνημόνιο για την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας. Είναι το θέμα της εξάρτησης της χώρας από τι αγωγέ ορυκτών καυσίμων πετρελαίου η ελλάδα όπω και οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν βαθιά κρίση σήμερα εξαρτώνται απόλυτα από εισαγωγέ πετρελαίου που κοστίζουν πολύ στην οικονομία του και συνεισφέρουν σε μεγάλο ποσοστό στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. μόνο για την περιοχή των μη διασυνδεμένων νησιών το κόστο εισαγωγή ετησίω πετρελαίου για να λειτουργούν οι μονάδε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. στο μνημόνιο λοιπόν θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην αποδοτικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων που θα μπορούσε να βελτιώσει και τα δημοσιονομικά της χώρας και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αναζωογονήσει την οικονομία. νομίζω λοιπόν ότι μια τέτοια πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ Σαλαβράκος Νικολάος. Κύριος Σαλαβράκος παρακαλώ. Σαϊνός. Ο κύριος Σαλαβράκος. Μπίνευ ούρ. Благодаря ви, господин председател. Колеги, имунитетът ми е потъпкан. Έχει προσβληθεί η ασυλία μου. Για ποιο λόγο. Εγώ την αλήθεια λέω, λέει ο κύριος Μπίνεφ. Υπάρχει μια πολιτική ένωση για την οποία ε, έχω εκφράσει κάποιες απόψεις. Η αστυνομία ήρθε, συνέλαβε κάποιους ανθρώπους, μεταξύ αυτών και εμένα, και με αντιμετώπισαν και ως κλιματή επειδή υποστήριξα την πολιτική ένωση αυτή, την ΓΚΟΡ. Και θα έλεγα ότι για την καταστολή είναι υπεύθυνο ο ίδιο ο, ίδιος ο Πρωθυπουργό. Βέβαια δεν τα κάνει ο ίδιο αυτά, αφήνει άλλου να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Η κυβέρνηση κλέβει από τους πολίτες, ε, καταπιέζει τους αντιφρονούντες. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Θα μπορούσε να στοιχίσει αυτή η στάση και ολόκληρες ε, και ανθρώπινες ζωές. Καλό λοιπόν να ληφθεί άμεσα δράση. Διότι αν οι Βρυξέλλες δεν μας προστατεύσουν από τη δικτατορία Πού πρέπει να πάμε, πρέπει να ζητήσω άσυλο, πού να πάω, να πάω στη Μόσχα, να πάω στο Πεκίνο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σήμερα στη Βουλγαρία, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη τώρα έχει το λόγο. The Η συνθήκη για την δημοσιονομική σταθερότητα θα τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ιρλανδία την 31η Μαϊδράτο με τι ευκαιρίε για να καταγγείλω την αντιδημοκρατική φύση τη όλη συζήτηση. Υπάρχει στρέβλωση τη δημοκρατική διαδικασία. που λέει ότι θα πρέπει να έχουν ε, ίδιο ε, χρόνο ε, ομιλίας, παρουσίαση στην τηλεόραση και οι δύο πλευρές. Και εκτός αυτού υπάρχουν και κάποια κεκτημένα συμφέροντα χωρίς καμία δημοκρατική εντολή. ένας ε, υποψήφιος ε, που και κατά το παρελθόν είχε λάβει πολύ ε, μεγάλο ποσοστό λόγου θα πάρει πάλι το λόγο, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μια αντίστοιχη εκστρατεία. Ο κύριος Γκότς, ένας οικονομολόγος, λέει ότι η Ιρλανδία παρέχει ασφαλές καταφύγιο, αποτελεί ένα φορολογικό παράδεισο. και διάφορα άλλα σχόλια. Μία πλατφόρμα του κυρίου Γκάντι, αντιδημοκρατική, την οποία θέλω να καταγγείλω. Ιδίω αν σα πω ότι οι 11 από του 12 βουλευτέ που είναι, δηλαδή βουλευτέ που είναι υπέρ του δημοσφίσματο, του ναι, μάλλον αγνοούνται. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία Κοπά έχει το Οι εκλογές στις 17 Ιουνίου θα είναι για την Ελλάδα οι πιο κρίσιμες μεταπολεμικά. Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν αν θέλουν μια κυβέρνηση υπεύθυνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση ή υποκύπτουν στο λαϊκισμό και στις εύκολες υποσχέσεις. Σε ένα τόσο κρίσιμο πλαίσιο, όπου τα διλήμματα τίθενται με δραματικό τρόπο, οι παρεμβάσεις από το εξωτερικό λειτουργούν αρνητικά, πυροδοτώντας αντιδράσεις ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν πρόσφατο παράδειγμα η πρόταση της κυρίας μέρκελ προς την ελληνική πολιτική ηγεσία για διεξαγωγή δημοψηφίσματος ναι ή όχι στο ευρώ την ίδια μέρα με τις εκλογές. η άποψη αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου γιατί μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να προτείνει δημοψήφισμα γιατί δεν υπάρχει βουλή που μπορεί να το αποφασίσει μια και έχει διαλυθεί εν ώψη εκλογών και γιατί πουθενά δεν γίνονται δημοψηφίσματα επειδή το απαιτούν κάποιοι εταίροι γιατί όταν προτάθηκε από την κυβέρνηση του πασόκ κάποιου μήνε πριν και με πιο συγκεκριμένο ερώτημα αντιμετώπισε αρνητικές αντιδράσεις διεθνώς με πρώτη την αντίδραση τη κυρία μέρκελ. κάθε τέτοιου είδου παρέμβαση είναι απόλυτα αντιπαραγωγική αυτή τη στιγμή. καλούμε την επιτροπή και το συμβούλιο να απέχουν από κάθε ενέργεια που δίνει την εικόνα παρέμβαση στα εσωτερικά κυρίαρχη χώρα. η ελλάδα χρειάζεται μια ενιαία φωνή στήριξη από την ευρώπη και όχι υποδείξει και απειλέ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, ο κ. Κυρακάκης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, γίνεται εκτεταμένη συζήτηση τον τελευταίο καιρό για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ ή κάποιοι μιλούν ακόμη και για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούν δυστυχώς πολύ περισσότεροι, πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Με κίνδυνο να προκαλέσουν κρίση πριν ακόμη φτάσουμε στις εκλογές ε, του Ιουνίου. Μιλούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όχι απλώς τις οικονομικές αλλά και τις κοινωνικές και τις γεωπολιτικές συνέπειες μια τέτοιας υπόθεσης. Θα ήταν καλύτερο αντί να, χωρίζουμε την ψήφο των Ελλήνων σε φιλοευρωπαϊκή και αντιευρωπαϊκή να συνειδητοποιήσουμε ότι κατά βάση ήταν ψήφος αντίδρασης στο πολιτικό σύστημα που έφερε την Ελλάδα στο σημείο που την έφερε και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την παραγωγική Ελλάδα η οποία δεν αξίζει να έχει την τύχη την οποία, η οποία της επιφυλάσσεται. Τα τελευταία δύο χρόνια η διαχείριση η οποία έγινε ήταν προβληματική σε σχέση με την πραγματική παραγωγική Ελλάδα η ανεργία χτύπησε κυρίως τον ιδιωτικό τομέα και για το γεγονό αυτό υπάρχουν και ευθύνες από την ευρωπαϊκή πλευρά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σταλαβράκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την ισορροπία μεταξύ λιτότητος και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών καλούνται να βρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες υπό την πίεση του εκλογικού αποτελέσματος σε γαλλία και ελλάδα αλλά και υπό το ανήσυχο βλέπαν των αγορών. τα αυστηρά μέτρα λιτότητα συνεχίζουν να δημιουργούν νέους ανέργους και γενικότερα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή στο σύνολο της ευρωπαϊκής ένωσης. τα εκλογικά αποτελέσματα τοπικών ή εθνικών εκλογών ανά την ευρώπη σημειώνω ιταλία γερμανία γαλλία αντιπροσωπεύουν μια γενικευμένη αντίδραση στην πολιτική της αυστηρής λιτότητας. είναι βέβαιο ότι απαιτείται χαλάρωση του γερμανικού προτύπου δημοσιονομικής πειθαρχίας και άμεση ανάπτυξη της οικονομίας για εξισορρόπηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και διατήρηση της συνοχής τους που απειλείται απειλείται και το νόμισμα κύριε πρόεδρε. πρέπει να σεβόμαστε τα ανεκτά επίπεδα των ευρωπαίων πολιτών και βάσει της αρχής της αλληλεγγύης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πρέπει να εξετάσουμε μια πιο ρεαλιστική λήξη με την έκδοση ευρωομολόγων την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τράπεζας και την έκδοση νέου χρήματος κύριε πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Χαιρετίζω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Σε αυτά επαναλαμβάνεται η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λύση δύο κρατών και εκφράζεται ανησυχία ότι αυτή η λύση υπονομεύεται από τον επικισμό κατεδάφιση οικειών και άλλων υποδομών στην ούτω καλούμενη περιοχή Σύ. Την ίδια στιγμή διπλωμάτες στην περιοχή καταγγέλνουν ότι τουλάχιστον 62 υποδομές που περιλαμβάνουν δεξαμενές ίδρυυσης και υγειονομικά συστήματα που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της κατεδαφίστηκαν από το Ισραήλ το 2011 πέραν των εκατοντάδων οικειών αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει χρηματοδοτηθέντα από την ευρωπαϊκή ένωση έργα αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ. αυτή τη στιγμή 110 υποδομές έχουν παραλάβει διατάγματα κατεδάφισης από τις Ισραηλινές αρχές και κινδυνεύουν να σωριαστούν σε ρήπια από στιγμή σε στιγμή. Οι υποδομές αυτές και τα έργα που ήδη καταστράφηκαν έχουν αναγερθεί με τα ειστερήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Ερωτώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν για να προστατεύσουν τα έργα που οικοδομήθηκαν με χρήματα των ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κορτέ Λάστρα, κ. Κορτέ Λάστρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλο και περισσότερες ε, υποθέσεις αρπαγής ε, παιδιών ε, λαμβάνουν, υπόψη, λαμβάνουν χώρα στην Ισπανία. Πρόκειται για δίκτυα, για κυκλώματα στα οποία συμμετέχουν θρησκευτικέ οργανώσεις, γιατροί, νοσηλευτές, ε, ουσιαστικά παίρνουν τα παιδιά ε, πολιτικών κρατουμένων και τα πηγαίνουν σε οικογένειες, συντηρητικές οικογένειες. Και είναι ένα ιστορικό δράμα, μια ιστορική τραγωδία στερούν ε, τα παιδιά από τις μητέρες που δεν έχουν πόρους. Πριν ε, από ένα χρόνο άρχισε αυτό το κύκλωμα να βγαίνει στο φως χάρη ε, στους ίδιους τους, στα ίδια τα θύματα, τους γονείς οι οποίοι πλέον έχουν μιλήσει γι' αυτό και απαιτώ να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει την, ε, τον αγώνα της ε, κατά της σωματεμπορίας και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί πατέρες και πολλοί μητέρες δυστυχώς δεν θα καταφέρουν να ξαναβρούν τα παιδιά τους. Είναι μια τραγωδία. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπρόντς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το να προσώσουμε μια χώρα που το χρέο προσπαθώντα να νίξουμε την, το λαό του σε, σε ανεργία και διαφέρει πολύ από τη 19ο αιώνα και την πολιτική τη Βρετανία που τελικά έχω να του πάτε στη φυλακή όμως να δανείζονται περισσότερο για να καλύπτεται η ζήτηση δεν θα μειώσει το χρέος. Ποσοτική ανακούφιση θα αυξήσει τη γενική ζήτηση χωρίς να αυξάσει την, το χρέος. Αλλά δεν αυξηθεί η παραγωγή, τελικά είναι πληθωριστική αυτή η τάση. Ποια πρέπει να είναι η αρχή. Ό,τι είναι φυσικός εφικτό θα πρέπει να είναι και οικονομικός εφικτό. Εάν έχουμε υποδομές και δουλειά που πρέπει να γίνει στις υποδομές και έχουμε εργάτε, οικοδόμου που είναι άνεργοι, αυτοί θα πρέπει να απασχοληθούν ούτω ώστε να κάνουν αυτό που χρειάζεται. Μπορεί να αποφευθεί ο πληθωρισμό, ναι. Εάν πλήρη πληρωμή για το έργο καθυστερήσει μέχρι να ολοκλήρωση του έργου, ε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να προσθεθεί στα αγαθά και υπηρεσίε. Η δημιουργία χρημάτων αυτόν τον τρόπο δεν είναι πληθωριστικό αν ταιριάζει χρονικά και ποσοτικά από αύξηση στα αγαθά και τι υπηρεσίε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφε Κουλιέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει και ε, λοιπόν, έχουμε την Πρωτομαγιά, γιορτάσαμε ε, την ημέρα της εργατιάς, ε, τα επιτεύγματα των εργαζομένων. Λόγω της οικονομικής κρίσης όμως απειλούνται αυτά τα δικαιώματα που οι κυβερνήσεις που δεν έχουν κοινωνική συνείδηση επιβάλλουν μέτρα λιτότητας και οικονομική πειθαρχία, δημοσιονομική πειθαρχία, αγνώντας όμως το μεγάλο βάρος που βαρύνει τους ώμους των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η οικονομική και χρηματοστική κρίση έγινε και κοινωνική κρίση. Θα πρέπει να ακούσουμε του εργαζομένου, θα πρέπει να είμαστε εμεί η φωνή των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη περιμένουν περισσότερα, περισσότερε δυνατότητε να απασχοληθούν, αυξήσει των επενδύσεων και δράσει που τονώνουν τι δυνατότητε απασχόληση για του νέου στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα δικαιώματά του. Η ανεργία στην Ευρώπη έφτασε ε, ρεκόρ 15 ετία. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι άνεργοι. Τα μέτρα λιτότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία που επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα τη ανεργία. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ προωθώ και υποστηρίζω την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εγγύηση που πρέπει να δίνονται στου νέου Ευρώπη, προστασία των δικαιωμάτων του. Κάθε νέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εργαστεί. Θα μπορεί να υποστεί κατάρτιση, συμπληρωματική κατάρτιση και να βρίσκει δουλειά μετά από τέσσερι μήνε στην ανεργία. Σε αυτή την πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Συνάδελφε Όσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 17 Ιουνίου ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Θα αποφασίσει για το μέλλον του, για τη μελλοντική του ζωή. Θα κάνει επιλογές ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο ο κύριος Τρισέ ε, που είπε αυτά που είπε στη συνάντηση της ομάδας των 8. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι θα πρέπει ο λαός να χάσει τελικά τη δικαίωμα της ε, ψήφου. Μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση που λέει όχι στη λιτότητα θα πρέπει να αντικαθίσταται από μια ομάδα επιτρόπων των Βρυξελών. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, όπως και η προσπάθεια ε, απειλής που στέφτε κατά τη ε, Ελλάδας. Η Ευρώπη είναι η αλληλεγγύη, η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται να γίνεται φτωχό ένα λαό ούτε να εκβιάζετε. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτείτε, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Διερωτηθείτε, «Ε, μπορείτε να δεχόσαστε τέτοια απεικιοκρατία, τέτοιου είδου απεικιοκρατική προσέγγιση όσον αφορά του Ευρωπαίου πολίτε. Είμαι σίγουρα ότι θα ζητήσουν τη δημοκρατία οι άνθρωποι τελικά. Σε ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Συνάδελφε ε, Τούντορ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάθε μέρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πράγματα που μας ε, δημιουργούν πραγματικό σοκ. Ε, άνθρωποι που τους δαγκώνουν ε, άγριοι σκύλοι. Υπάρχει το περιστατικό αυτού που ήταν σε απομόνωση στην Ιταλία και που ήταν αντικείμενο ξυλοδαρμών και στη συνέχεια των αγνόησαν και πέθανε μετά από μακρά απεργία πείνας. Όλα αυτά είναι περιστατικά απάνθρωπης μεταχείρισης. όπως απάνθρωπη μεταχείριση επιφυλάσσουμε και στους ε, αγωνιζόμενους για την ειρήνη, στους ακτιβιστές της ειρήνης. Βλέπουμε ότι ε, άνθρωποι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, παιδιά με ένα λουλούδι στο χέρι που μάχονται για την ειρήνη αντιμετωπίζονται με βία μέσα και τους ε, κλωτσάνε και τους ε, σπρώχνουν. Υπάρχουν πολίτες που προσπαθούν να αμυνθούν. Ο Χίτλερ δεν έχει πεθάνει. Ο Χίτλερ ζει με άλλη μορφή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Παπαδοπούλου και δημοκρατικέ εκλογέ στη Γαλλία, Φιλανδία, Ολλανδία και Ελλάδα έχουν καταδείξει την αυξημένη διαμαρτυρία των πολιτών ενάντια στην αυστηρή λιτότητα και τι αποτυχεμένες συνταγέ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο νέος αέρας αλλαγής στη Γαλλία και γενικότερα αναζωογονεί την ελπίδα πώς θα τερματιστούν επιτέλους οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και πώς η Ευρώπη θα ξαναμπεί στη λογική της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της πραγματικής κοινωνικής αλληλεγγύης εύχομαι η ελλάδα να αποκτήσει σύντομα στι 17 ιουνίου κυβέρνηση και να παραμείνει στο ευρώ γιατί τυχόν αποχώρησή τη θα έχει αρνητικέ αλυσιδωτέ επιπτώσει στι χώρε του ευρωπαϊκού νότου στην ευρωζώνη και στη συστημική σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματο. οι ομοί εκβιασμοί τη κυρία μέρκελ και άλλων αξιωματούχων σε βάρο του ελληνικού λαού είναι επικώς απαράδεκτοι και αχρίαστοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε, ο κ. Φεραίρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις τελευταίες τελευταίες εβδομάδες στην Πορτογαλία είδαμε να πηγαίνουν προς τα πίσω όσον αφορά την οικονομία της, τα πολιτιστικά της, οι παρεμβάσεις του Δούνου του και οι επιθέσεις κατά εκείνων οι οποίοι προσπαθούν να σταματήσουν την κυβέρνηση από την εφαρμογή των μέτρων που θέλει να επιβάλλει, που είναι επίθεση στο λαό της Πορτογαλίας. Άλλη μια επίθεση κατά μια ίδια δύναμης δημοκρατίας είναι αυτή. Η, η διακοπή των αυξήσεων, η μείωση των διακοπών, η απώλεια όλων των δικαιωμάτων εργαζομένων, η υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων, Όλα αυτά, εκατομμύρια επί εκατομμυρίων ευρώ, θα βγουν από τα χέρια, φύγουν τα χέρια των Πορτογάλων εργαζομένων, θα χαθούν πολλές θέσει εργασίας. Και αυτό μια εποχή που η ενεργεία ήδη είναι σε ιστορικά ύψη. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα, και το επαναλαμβάνω αυτό, απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες που θα διαδηλώνουν στην ε, Λισαβόνα να πούν ότι αρκετά πια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις του ενός λεπτού και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκθεση Ρίτα Μπορσελίνου σαν στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής